μέσα σε 24 ώρες υπάρξει μια αίτηση από μια πολιτική ομάδα ή 40 μέλη του Κοινοβουλίου θα τεθεί η γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής σε ψηφοφορία. Αλλιώς θα θεωρηθούν